Hello. Uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να λάβετε τις θέσεις για να αρχίσουμε αμέσως τη συνεδρίασή μας. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam Αρχίζει και πάλι η συνεδρίασή μας που διεκόπη στις 9 Σεπτεμβρίου του 2010. Και με μεγάλη λύπη μου πρέπει να σας ανακοινώσω τον θάνατο του Έγκον Κλέψου που ήταν το 80, 90, το 1992-1994 πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κλέψου είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ε, ζωής του στο ευρωπαϊκό όραμα. Ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για πέντε θητείες επί 20 χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να ποτίσουμε φόρο τιμής στον κύριο Κλέψου, τηρώντας ενός λεπτού υγιής. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι το βιβλίο συλληπιτηρίων έχει ανοίξει και μπορείτε να το υπογράψετε. Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, πολλά συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ότι την ερχόμενη 5η 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει γενική απεργία στη Γαλλία. Αυτή η συνδικαλιστική δράση θα καλύψει τις ε, ε, μεταφορές, θα ξεκινήσει ε, η απεργία στη Δετάρτη στις 8 το βράδυ και ενημερωθήκαμε επίσης ότι η απεργία πιθανώς να ξεκινήσει και πιο νωρίς πριν από τα μεσάνυχτα, γύρω στις 20 όπω σα είπα. Και η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε ωστόσο ότι το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει τις εργασίες του και θα λήξει η συνεδρίαση την Πέμπτη μετά τις ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά τι πτήσει και τα τρένα, θα επηρεαστούν πιθανότατα από την απεργία, όπως και οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες Γι' αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για όλους